I Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ, γιατί πολλοί από τους βουλευτές μας θέλουν ακόμα να φύγουν σήμερα από τις Βρυξέλλες, να πάρουν τα τρένα τους, τα αεροπλάνα τους. Οπότε πρέπει να δουλέψουμε αποτελεσματικά, γρήγορα. Και θα το κάνουμε. Έχουμε πολλές ψηφοφορίες μπροστά μας. Και μετά από την ψηφοφορία θα έχουμε και μια σύντομη και πολύ αποτελεσματική συνεδρίαση των συντονιστών. Οι συντονιστές λοιπόν να παραμείνουν παρακαλώ. Και όσοι είναι να φύγουν, θα φύγουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αρχίζουμε λοιπόν την ψηφοφορία. πρώτο θέμα για προφορική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφορική ερώτηση όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ψηφίζουμε. Συμβαστικό κείμενο. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Ερώτηση 4 τώρα. Πάλι συμβιβαστικό κείμενο. Με μια προφορική τροπολογία της κυρίας Χάρκιν. Προσθέτει τη λέξη εθελοντική. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ελέγχουμε μια την προφορική αυτή τροπολογία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 26 ψήφοι υπέρ. Ερώτηση 5. Πάλι έχουμε συμβαστικό κείμενο. Η κυρία Γκέριους έχει το λόγο. Συγγνώμη, συγγνώμη που σας καθυστερώ. Αλλά δεν υπάρχουν κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την ερώτηση 5 για την εταιρική ευθύνη για τις πληροφορίες και την ενημέρωση δηλαδή και τη διαβούλευση με τους εργαζόμενους. Όπως ίσως θα θυμόσαστε, η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία εγκρίθηκε ήδη από το 2013 στην Ολομέλεια και αντιληφθήκαμε ότι το κείμενο της ερώτησης 5 δεν ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το κείμενο που εγκρίναμε τότε. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω μια προφορική τροποποίηση στην ερώτηση 5 που να λέμε θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια νομική πράξη, όχι νομικό πλαίσιο, αλλά νομική πράξη για ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζόμενους σε περίπτωση που υπάρχει η αναδιάρθρωση, έτσι όπως κτλ. κτλ. Για να το ευθυγραμμίσουμε δηλαδή με την αρχική πρόταση. Πρόεδρος, καλώς. Ψηφίζουμε λοιπόν το συμβαστικό κείμενο στην ερώτηση 5 με την τροποποίηση. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίστε. Από το ΕΛΚ ψηφίζει ένας παραπάνω. Τώρα εντάξει. Καλώς. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. Τώρα την τροποποιημένη ερώτηση ψηφίζουμε υπέρ παρακαλώ. Α, συγγνώμη λέει πρόεδρος, βέβαια ηλεκτρονικά πρέπει να ψηφίσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεν θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Ωραία, συνεχίζουμε. Ψηφίζουμε τώρα για το κοινωνικό dumping στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροπολογία 1 είναι μη αποδεκτή. Οπότε περνάμε στην τροπολογία 142. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 143. Υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται νομίζω, αλλά θα ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορίας. Α, πάλι από το ΕΛΚ. Ψηφίζει ένας παραπάνω. Εντάξει τώρα. Εγκρίθηκε με δύο ψήφους διαφορά. Συ... 145 τροπολογία, 146 και 147 μαζί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική α. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική β. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική B, A. Υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 187 και 188 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική γάμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική CA γάμα Α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σελίδα 11 τώρα. 215 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 219 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας, τσίμα τσίμα, ισοψηφία. 220 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική D δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 232 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική DA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 234 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία ε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γυναικών 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική F. Α, όχι, προηγουμένως οι 245, 46, 47, 48. Υπέρ παρακαλώ αυτών των τεσσάρων κατά αποχές απορρίπτονται. Τώρα πάμε στη συμβαστική F. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 18 πάμε τώρα για την τροπολογία 278 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 279 και 280 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη σελίδα 20. Έχουμε την τροπολογία 293. Και 204, 205, 206, 207, 298. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική H υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Επόμενη σελίδα 21, τροπολογία 307. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πιστεύω, αλλά θα ελέγξουμε καλύτερα για την 307. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα της φοφορίας, απορρίφθηκε. Τροπολογία 310. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 313 υπέρ, κατά, 313 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 315 με 316 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική ΑΙ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J, J υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 24 τώρα και μετά τροπολογία 346 και οι επόμενες υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτονται συμβαστική κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω, αλλά σε ελέγξουμε. Είδα κάποια βεβαιότητα στον τρόπο με τον οποίο ψηφίσατε. Πέρα στις προφορίες, ναι, εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Ε, δεν σηκώσατε τα χέρια σας, τι να κάνω, λέει η Πρόεδρος. Τροπολογία 358 τώρα. και οι υπόλοιπε μέχρι και 362 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβαστική L υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σελίδα 29 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σελίδα 31 τώρα. 4.14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4.15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε θέλετε. Εντάξει, 415 ελέγχουμε ηλεκτρονικά, ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Σελίδα 32, τροπολογία 420 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε για την 420. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 423 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία δεν θέλετε να ελέγξουμε. Ήταν σαφές. Ωραία. 425 τώρα. 426 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 425 και 426. Ωραία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για να ελέγξουμε. Πέρα τη υποφορία. απορρίφθηκαν. Τροπολογία τραν 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική R. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τραν 18. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 444 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τραν 21. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τραν 20. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 462. Αλλά όχι, συγγνώμη, λέει πρόεδρος, καταπίπτει. Τροπολογία 464 τώρα. Α, και αυτή καταπίπτει, διορθώνει πρόεδρος. 465 και 466 τότε μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβαστική π υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 480, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 481, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία, για την 481 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρα στις φοφορίες. Απορρίφθηκε. Τραν 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τραν Α, όχι. Πάμε στη σελίδα 39. Κύριε Πρόεδρε. Μία παράκληση. Όλα πολύ ωραία τα κάνετε. Όμως όλοι έχουμε, καθώς φαίνεται, διαφορετικούς καταλόγους πλήρω ε, ψηφοφορίας. Άλλος είναι στη σελίδα 39, άλλος στη σελίδα 43. Ε, θα μπερδευτούμε. Είναι περίπλοκο το θέμα. Πρέπει να προσέξουμε για να μην κάνουμε λάθος στην ψηφοφορία. Ναι, γνωρίζω ότι κάθε ομάδα έχει τη δικιά της ομάδα. Εγώ έχω τον κοινό κατάλογο που είναι για όλους μας. Εντάξει, δεν θα λέω σε ποια σελίδα είμαστε, αφού προτιμάτε. Εντάξει, για να μην σας μπερδεύω. Λοιπόν, τώρα που ήμασταν. Είμαστε στις τροπολογίες τραν 16 και τραν 19, που τις ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Νομίζω, αλλά εντάξει, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε λοιπόν. Πέρα της φοφορίας Εγκρίθηκε. Εντάξει, έκανα λάθος. Τροπολογία 503. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 504. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ωραία. 504. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της φοφορίας. Τραν 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 507. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ωραία, για την 507. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα της φοφορίας. Ισοψηφία πάλι. Τραν 26, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τραν 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 523. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 524. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 525. Υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία. 525. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη φοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 528. 529 και 530 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβαστική S. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική S, α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 539. Μαζί με την 540, 541, 542, 543, 544 και 545. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβαστική ταφ α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική ταφ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 564 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σύμβιβασ... Όχι, 565 πρώτα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Α, όχι, απορρίπτεται, διορθώνει η πρόεδρος. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Ε, συμβαστική βή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ΒΑ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τραν, όχι, 586 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 584 υπέρ, κατά, αποχές, Θα ελέγξουμε. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρασε της πληροφορίας εγκρίθηκε. Συμβαστική W. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 587, 588, 589 και 590 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβαστική X, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γυναικών 9, φάμε 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 604, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ωραία. 604 τροπολογία ηλεκτρονικά πέρα της φοφορίας Απορρίφθηκε. Τροπολογία 607. Υπέρ, κατά, αποχές, ξανά. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 608 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. 608. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. Εγκρίθηκε. Με 27 υπέρ. 609 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τα ελέγξουμε. 609 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 29 ψήφι υπέρ. Τροπολογία. Συμβαστική μα. Α, όχι. 610 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Y. Y. Y υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 623, 624 και 625 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Z, Z υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 647 τώρα. Υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε. 647 λοιπόν ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα τη φοφορία. Ισοψηφία. 649 και 650 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβαστική ΑΑ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 666 μαζί με την 667, 668, 669 και 670 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβαστική ΒΒ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΚΑΠΑ Α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γυναικών 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική σι γάμα γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 687 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Α, θα ελέγξουμε. 687, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. Απορρίφθηκε. 688 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Νομίζω θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για την 688 ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. Ισοψηφία. 690, 691, 692, 93, 94, 95 και 696 μαζί υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική DD υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 701, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. να ελέγξουμε. 701, ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της φοφορίας. Απορρίφθηκε πράγματι. Τώρα τροπολογία 702. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Όλο το κείμενο χωρίς τις λέξεις in the worker mobility package, το πακέτο κινητικότητας ε, εργαζόμενων. Και στο δεύτερο ψηφίζουμε μόνο αυτές τις λέξεις. Λοιπόν, το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία. 703. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε για την 703. Πέρας της φοφορίας. Εγκρίθηκε. Ερχόμαστε στις αιτιολογικές αναφορές. Τροπολογίες 2 και 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Καταπίπτει 4. 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 7 καταπίπτει, 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, να ελέγξουμε για την τροπολογία 9 λέτε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 9. Ψηφίστε. Πέρα τη φοφορίας.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 αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Αλλά να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά για την τροπολογία 23. Ψηφίστε. Πέρα της φοφορίας. Απορρίφθηκε. Τραν F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Τραν F. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Τραν F. Ψηφίστε. Πέρας της φοφορία απορρίφθηκε. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα ελέγξουμε για την 25. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, θα ελέγξουμε για να μην καθυστερούμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 27. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική AC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Γυναικών Β υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46. Υπέρ. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική. ΑΕ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γυναικών δέλτα D υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Γυναικών ε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 50 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, having regard as ε, features. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Από such as έως transport. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρας της φοφορίας. Απορρίφθηκε. Τραν α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τραν Β, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 107, υπέρ. Κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 107. Ψηφίστε. Πέρασε φοφορίας. Εγκρίθηκε. 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, Θα ελέγξουμε για την 55 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. πέρα τη ψηφοφορίες... Απορρίφθηκε. Συμβαστική AG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική μείον α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική H. υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 74. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 75 πέντε υπέρ, κατά, αποχές, δεν σηκώνετε τα χέρια σας, οπότε δεν βλέπω πώς ψηφίζετε και θα ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Για μια στιγμή. Να δούμε μήπως έχει ήδη εγκριθεί και καταπίπτει. Α, ναι. Εντάξει. Καταπίπτει. Έτσι λέει η Αντιπρόεδρος. Οπότε πάμε στην τροπολογία 76. Υπέρ. Α, όχι, διορθώνει η πρόεδρος. Ωραία. Τροπολογία 85, υπέρ. Μαζί με την 86. Ε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Νομίζω να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική ΑΙ. Υπέρ. ΑΙ. Διακοπές χρειάζομαι, λέει ο Πρόεδρος. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 89 και 90 μαζί υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Α, να ελέγξουμε πρώτα. Ωραία. Για την 89 και 90 ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα της φοφορίας απορρίφθηκαν. Συμβαστική AJ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AL. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 108. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 110. Με προφορική αλλαγή από τον εισηγητή, το 0,6% να γίνει 0,7%. Με την προφορική λοιπόν αλλαγή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 111. Πάλι έχουμε και εδώ μια προφορική τροποποίηση. Με την προφορική τροποποίηση λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκατόν υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. 122 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 123 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ελέγχουμε για την 124 ηλεκτρονικά ψηφίστε. Πέρας της φοφορίας. Απορρίφθηκε. Με δύο ψήφους διαφορά. 126 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 130. Ψηφίστε. Πέρας της φοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική ΑΚ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και φτάσαμε στο τέλος αυτής της ψηφοφορίας. Τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 37 ψήφοι υπέρ, 7 κατά. The roll call vote result will be in... Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ευχαριστώ και τους κοιόδης. Ξέρω ότι είχατε 20 συναντήσεις και οδόν. Τεράστιος ο ρυθμός. Για το βραβείο Γκίνες. We proceed now with the draft report by Mr. Να προχωρήσουμε με το σχέδιο έξιση του κυρίου Κρασινοντέμσκι. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε για την 59. Άρχισε την ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 61 ε, καταπληκτή. 65 μαζί με την 66 έχουν αποσυρθεί, οπότε πάμε στη συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα ξαναπάμε στη συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβεστική 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ελέγχουμε για την 103. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 113. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Budget 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρετζι 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Budget 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 333 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Ρέτζι 3 υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. Budget 1 υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Budget 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Reggie 4 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Budget 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Α, α καταπίπτουν. Ρέτζι 9. Υπέρ. Κατά. Για τη Ρέτζι 9. Υπέρ. Ρέτζι 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129. Υπέρ. Με προφορική τροπολογία με συγχωρείτε που φορεί και τροπολογία. Ναι, είπα ερώτηση, θα μια φορά είναι ερωτήσει. Ορολογία που ζήτησαν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική επτά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική το υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...88 με προφορική τροπολογία από τον κύριο Πάβελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 148 με προφορική τροπολογία από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 149 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, απορρίπτεται συγγνώμη, 160 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 159 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 161 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 293 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκατόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ κατά εγκρίνεται. 196 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 196. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Α, 197 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 206 μαζί με την 207 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 208 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 209 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 256. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 248. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Ελέγχουμε για 248. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα. Εγκρίνεται. 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 233 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 234 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 200... 239 έχει αποσυρθεί, 16. συμβαστική 16 υπέρ, κατά, εποχές, Νομίζω 251 τώρα, υπέρ, κατά, εποχές, Εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεν ήταν παρατήρηση. Ωραία. Ρέτζι 19. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μπάτζετ 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. «352 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται». Όχι, έχει καταπέσει. Ρέτζε 2 και αυτή έχει καταπέσει. 263 υπέρ κατά αποχές θα μπορούσε να, απορριφθεί, να απορριφθεί, αλλά πρέπει να το ελέγξουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Ναι, ναι, απορρίφθηκε. 264 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 265. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Σύμβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. 287 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 288 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 289 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 290 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε για την 290 90 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 292 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 304 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 305 έλεγχος για το 304 να ελέγξουμε η ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται πέρας απορρίβεται. 305 και 306 μαζί. Να μην πω τώρα ότι έρχεται η ψηφοφορία υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε για την 305 και 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αγκρίνεται. 307 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεστή 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 311 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 312 υπέρ κατά αποχές 313 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 314 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 317 υπέρ κατά αποχές πρέπει να γίνει έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία 317 πέρας αυτής είναι ένας υπεραριθμός στα μέλη των σοσιαλιστών. Απορρίπτεται. Συμβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 332 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 325 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 326 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 327 3-3-4, 334 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 335, 335 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 336 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 337 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 338 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 339 υπέρ κατά αποχές απολύτω 340 υπέρ κατά αποχές απολύτω 341 υπέρ Κάνουμε έλεγχο για την 340. Άρχεται η ψηφοφορία. 340. Εγκρίθηκε με 31 ψήφους, 341. Ψηφίζουμε την 341 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 342 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 343 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 345, 345 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 246 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 347 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος για την 347. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με 31 ψήφους, 348 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 350. 350 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 351 υπέρ, κατά, θα μπορούσε και να απορρίπτεται, αλλά ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. 351. Πέρας. Απορρίπτεται. Budget 8. Καταπίπτει. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ψηφίσουμε ξανά με τα χέρια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. 353. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 354. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 300. 55, την ψηφίζουμε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 357, υπέρ, κατά, αποχές, Έλεγχος για τον 357. Πέρας. απορρίβεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Αιτιολογική σκέψη α και το τοπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία για να είμαστε βέβαιοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μεγάλη ψηφία. Με 13, those in favor, those against, abstentions carried. Uh, budget C, those in favor, those against, abstentions carried. Amendment 14, those in favor, those against, abstentions carried.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 Uh, Amendment 20, those in favor, against, abstentions carried. Amendment 21, those in favor, against, abstentions carried. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποθέσεις, εγκρίνεται. 33 με κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποθέσεις, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποθέσεις, Έλεγχο για το δεύτερο τμήμα της 33 άρχεται η ψηφοφορία πέρασε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 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα έλεγα έλεγχος, έλεγχος για την τροπολογία 6 άρχεται η ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται. επτά υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε για το σύνολο της έκθεσης ως τροποποιήθηκε. Βάσει το πρωτοκόλλο. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρα της ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ. Καλή ψηφοφορία. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή και όλους τους κοιόδης για όλη τους τη δουλειά. Now we vote on the draft report. Τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης της Λαούρα Αγκαία. Συμβιβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται. Πέρας. 39 ψήφι υπέρ, 5 κατά. Τώρα, Περνάμε στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικά θα ψηφίζουμε. Πέρας. Η ψηφοφορία θα συμπεριληφθεί στην έκθεση. 40 ψήφοι υπέρ, κατά. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Την ευχαριστούμε πολύ, καθώς και όλους τους κοιόδης. Ψηφίζουμε τώρα μία ψηφοφορία για την έκθεση Σόγκορ για την τριμερή κοινωνική συνοδό κορυφής για την ανάπτυξη και απασχόληση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 50 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Καταπληκτικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ όσοι εργαστήκατε για την έκθεση αυτή. Τώρα, περνάμε στη δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Έχετε τον κατάλογο. Θα αρχίσουμε με την συμβαστική ΑΑ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 11. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 15. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά, αν και νομίζω πως απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 16. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε και το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 25 και 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. Συμβιβαστική ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε την συμβιβαστική ε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. μυστικές πληροφορίες συζητάμε. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Τροπολογία 28. Πέρας ψηφοφορίας για την 28 απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος, τροπολογία 29. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Δεν διαφωνείτε, βλέπω. Θέλετε να ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε, λοιπόν. Τροπολογία... Όχι, περνάμε στην τροπολογία 32. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Λοιπόν, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 31. Μας ζητήθηκε. ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 31. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Κατά τμήματα. Πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 17. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 17 του κυρίου Μέσεριτς. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ελέγχουμε και ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37 καλύπτεται από τον 36. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 39. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Όχι. Τροπολογία 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 48. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική F. Όχι, με συγχωρείτε, λέει η πρόεδρος. Συμβιβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε την συμβιβαστική F. Θα την ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 42. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41. Ψηφίζουμε την τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 43. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Συμβιβαστική G. Όχι. G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 55. Άρχεται. Πέρας. Τροπολογία 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική H. Ήτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε την συμβιβαστική H. Ήτα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Μάλιστα. Είμαστε χωρισμένοι, βλέπω. Τροπολογία 57. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Θα ελέγξουμε την 57. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Τροπολογία 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 62. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66. Υπέρ. Όχι καταπίπτει, λέει πρόεδρος. Περνάμε στην συμβιβαστική γιώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την συμβιβαστική γιώτα. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβιβαστική Ι. Πέρας. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο παραπάνω. Τροπολογία 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 68. Άρχεται. πέρασε, Απορρίπτεται. Τροπολογία 69. Μαζί με την 70, 71 και 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 μαζί με την... Όχι, μόνη της. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική J, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη συμβιβαστική J, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 79 και 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβιβαστική κάπα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά συμβιβαστική κάπα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 90. 2. Προφορική τροπολογία της κυρίας Τρεμπέζιους. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 94. Προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 95. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 97. Περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί ηλεκτρονικά. εισηγητής. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι θα καταψηφίσω την τροπολογία. Την έκθεση. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Λυκιώτης. Θα ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα λοιπόν θα καταγραφεί στα πρακτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Μας μπέρδεψε κάπως η σημερινή ψηφοφορία. Και αυτό σημαίνει πως πραγματικά χρειαζόμαστε διακοπές. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για αυτό το ε, καλοκαίρι που έρχεται λίγο νωρίτερα μια που τελειώσαμε νωρίτερα. Θα τα ξαναπούμε 31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου στις επόμενες συνεδριάσεις μας. Τώρα ήρθε η ώρα για τους συντονιστές.